People Όλοι είναι διάθετοι σήμερα το πρωί. Το καταγράφω λοιπόν με μεγάλη ευχαρίστηση αυτό. Θα μπορούσατε όμως όλες αυτές τις συζητήσεις να τις κάνετε λίγο αργότερα προκειμένου να καλύψουμε και όλα τα σημεία της μερίσιας διάταξης. Σας περάσουμε στο πρώτο σημείο, σχέδιο μερίσιας διάταξης. Πρέπει να σα πω ότι πρόκειται για την τέταρτη συνεδρίαση που γίνεται από κοινού με την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων όσον αφορά την διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εδώ τη σχετική στρατηγική έρευνα τη Ευρωπαϊκή Μεσολαβήτριας. Αυτή είναι η μόνη ανακοίνωση που είχα να κάνω. έχει διανεμηθεί το σχέδιο σα διάταξη έχει διανεμηθεί στα μέλη και των δύο επιτροπών, και τη δικιά μα και τη Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων. Μπορούμε να εγκρίνουμε τη μερίσια διάταξη. Πολύ ωραία. Καμία αντίρρηση. Ας περάσουμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 24 η Σεπτεμβρίου. Μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, έτσι δεν είναι πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε ευθύ αμέσως με την ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε μαζί σας τις κάρτες, να τις έχετε βάλει στο μηχάνημα, στη συσκευή. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την κοινή έκθεση σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γιώ Λάινεν είναι ο εισηγητής, είναι εδώ, είναι μαζί μας, μάλλον καθοδόν. Και για να τούμε επίση είναι η συγγήτρια, η οποία όμω είναι παρούσα από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Μάλλον λάθο. Συμβαστική 5. Λέει πρόεδρο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Διορθώνει πρόεδρο. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 41. Υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 42 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα, μάλλον η 11 έχει αποσυρθεί, στην 51 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση για ποια τροπολογία, για την 56. Πολύ ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την τροπολογία 56. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Ψηφίζουμε τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πίτερ, ψηφίζεις υπέρ των πάντων σήμερα. Πολύ ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. Λυπάμαι, Πίτερ. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 75. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77, η τροπολογία αυτή είχε αποσυρθεί, άρα πάμε στην συμβασική τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία 15 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, η συμβαστική 15 εγκρίθηκε είπαμε. Περνάμε στην τροπολογία 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές Ας ε, ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 92, άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας το επαληθεύσουμε. Θα πρέπει να σηκώνετε το χέρι σας για να βλέπω καλύτερα. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 92, η οποία εγκρίνεται, αλλά πραγματικά πρέπει να σηκώνετε το χέρι σας. Όταν λέω ότι νομίζω ότι εγκρίνεται, το λέω επειδή ελάχιστα χέρια σηκώνονται. Λοιπόν, 93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Λοιπόν, πολύ καλή πρωινή άσκηση αυτή να αλλάζετε και τα χέρια από εκεί που 100 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του σχεδίου έκθεσης ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Δείτε το αποτέλεσμα, καταπληκτικό, πολύ θετικό. Συγχαρητήρια στους δύο συγητές μας. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την εξαιρετική συνεργασία. Now, τώρα. Δεν τελειώσαμε αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ολοκληρώσαμε. Ας ακούσουμε τώρα τι έχει να πει η Ντανούτα, η επικεφαλής Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ των δύο επιτροπών μας. Ισχύει ότι ποτέ δεν συμμετείχα σε μια ε, κοινή ε, συνεδρίαση όπου η Προεδρία της ΑΦΚΟ δεν συμμετέχει σε όλη την διαδικασία. Το σημαντικό βέβαια είναι το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι όταν δύο ε, επιτροπές ε, εργάζονται υπό, την, υπό το άρθρο 55, δεν είναι και ότι το πιο ομαλό, όμως επειδή το ζήτημα ήταν τόσο σημαντικό, μας ένωσε τις δύο επιτροπές μας, αλλά και ένωσε τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Αν θυμάστε καλά την πρώτη κοινή συνεδρίαση υπό την Αυστριακή Προεδρία, διότι ε, αναφερόμασταν κυρίως στο Συνοβούλιο είχαμε ένα πολύ θετικό μήνυμα από τους Αυστριακούς ούτως ώστε να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις ε, και ε, να ενημερώσουμε το Συμβούλιο ότι υπάρχει μεγάλος, υπήρχε μεγάλος χώρος βελτίωσης ε, ούτως ώστε μέχρι το τέλος της θητείας να αφήσουμε πίσω μας ένα μήνυμα σχετικά με το ότι τα με το ότι ε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι διαφανής ε, και αυτό θα βοηθούσε βέβαια και τους πολίτες να καταλάβουν καλύτερα το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που είχαμε αυτή τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και ελπίζω ότι στο μέλλον αν ξαναβρεθούμε η συνεργασία μας θα είναι, θα είναι τόσο παραδειγματική. Ευχαριστώ πολύ Τανούτα και ευχαριστώ και σε όλους. Οι Επιτροπές ε, Αναφορών ε, έκανε τον, ε, τη δουλειά της, δουλέψαμε καλά με την Επιτροπή ΑΦΚΟ και βοηθήσαμε στην δημιουργία καλής νομοθεσίας και η συνεργασία μας δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Ευχαριστώ λοιπόν όλους και τώρα λίγα λεπτάκια για να εγκαταλείψετε την αίθουσα όσοι δεν θα μείνετε και εύχομαι σε όλους μια πολύ καλή μέρα.